meine Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια μικρή καθυστέρηση. Πάντως, μπορούμε να αρχίσουμε τώρα νομίζω. Έχουμε λίγο χρόνο στη θέση μας. Κυρία Λίχτινμπεργκερ νομίζω ε, θέλει το λόγο για την ημερήσια διάταξη. Αμέσως κυρία Λιχτεμπέργκερ παρακαλώ. Κυρία Λιχτεμπέργκερ. Ναι, μια παράκληση γιατί αύριο στην Επιτροπή Μεταφορών έχουμε από τι 9 μέχρι τις 12.30 ψηφοφορίες με 2.000 τροπολογίες εν όλο. Και δεν θέλω να παρακαλέσω το θέμα των ε, ε κεφαλαίων του προϋπολογισμού να το δούμε σήμερα ή δυνατόν. Καλώ, λέει ο πρόεδρο. Ποιο σημείο ήταν αυτό τη ημερήσια διάταξη, να το κοιτάξουμε. Ναι, έχουμε αρκετό χρόνο, μπορούμε να το καταφέρουμε. Αρκεί να μου αποκαλύψετε ποιο ήταν αυτό. Ήταν η, η απαλλαγή του 22. Ή να το κάνουμε πριν από τις ε, απόρριτες συνεδριάσεις τις κλειστές μετά το 6α πριν το 7. Καλώς. Διορθώνουμε λοιπόν έτσι την σε διάταξη. Και έτσι, σήμερα, αφού μετά τις 6 και 10, μετά τον κύριο Αλμπερτίν και την ακρόαση, θα ασχοληθούμε με ένα μια πρόταση της ε, νομικής υπηρεσίας για ένα ζήτημα που αφορά προθεσμίας, προθεσμίες και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αύριο. Μετά την ψηφοφορία έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φώστερ στο σημείο 23, προστασία των ιδιωτών. Έχουμε το θέμα του κυρίου Μπερλίνγκουέρ για τα ευρωπαϊκά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που αύριο θα το δούμε μετά το σημείο 17 και έτσι αύριο έχουμε μία υπόθεση εκ από το, από το Βελγικό σταγματικό Δικαστήριο για την ασυλία του κυρίου Στάτλερ που όμως επειδή είναι ασθενής θα πρέπει να αναβληθεί είναι επαρκής η αιτιολόγηση και έτσι όπως είπαμε νωρίτερα το θέμα της κυρίας Λιχνιμπέρκερ έρχεται μετά το σημείο 6 στη μερική διάταξη. Αυτές ήταν οι αλλαγές. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης για να σας επισημάνω ότι έχουμε προσκληθεί ως μέλη της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων να λάβουμε μέρος ε, ε, στην εκδήλωση της κυρίας Ρέντινγκ που προβλέπεται αύριο απόγευμα να λάβει χώρα μετά τις 3 μαζί με την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών με θέμα το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Έτσι λοιπόν, μια και είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, καλό θα ήταν κάποιοι από εμά να πάνε εκεί. Και θέλω να επισημάνω επίσης ότι αύριο πρέπει να έχετε μαζί τις κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρακτικά. 6 Νοεμβρίου, 19 Νοεμβρίου, τα δύο πρακτικά που έχετε λάβει, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της ε, απόψινής συνεδριάσεως, εγκρίνονται. Και καλωσορίζω τον κύριο Λουκά, εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας, τον Υπουργό. Σήμερα έρχεται να μας μιλήσει για το τέλος, για τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας και έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να συζητήσουμε μαζί του. Σας καλωσορίζω καταρχάς, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε το έργο που έχει επιτελέσει η Κυπριακή Προεδρία κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2012. Η Κυπριακή Προεδρία κατά το εξάμεινο που πέρασε εστίασε τις προσπάθειές της στη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης που θα είναι πιο αποτελεσματική τόσο για τους πολίτες της όσο και για τους γείτονές της. Όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. Σε σχέση με τον τομέα αυτό θα αναφερθώ πρώτα στην αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 1 ο οποίος αποτελεί το θεμέλιο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικά θέματα. Ο κανονισμός καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και διευκολύνει την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη δική σας συνεργασία και στήριξη, συνεχίζοντας το επιτυχημένο έργο των προηγούμενων Προεδριών, κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό επί Κυπριακής Προεδρίας. Η πρόταση υιοθετήθηκε στο τελευταίο μας Συμβούλιο ΔΕΗ και ακολούθως στις 12 Δεκεμβρίου υπογράφηκε η υιοθέτηση του κανονισμού από τον Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα και από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σούλτς στο Στρασβούργο. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον εισηγητή κ. Τατέου Ζεύσκα για την εξαιρετική συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε επίσης γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο ΔΕΗ Δεκεμβρίου αναφορικά με την πρόταση κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις. Η συγκεκριμένη πρόταση κανονισμού είναι πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες και αποτέλεσε προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας με τη διεξαγωγή σημαντικού αριθμού συναντήσεων σε επίπεδο ομάδας εργασίας. Ο στόχος της πρότασης είναι η εγκαθίδρυση ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει ότι όλα τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε ένα κράτος μέλος θα εποφελούνται από ένα γρήγορο και αποδοτικό μηχανισμό αναγνώρισης εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ελεύθερη κυκλοφορία των μέτρων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή αποτελεί την τελευταία εκκρεμότητα του νομοθετικού πακέτου, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπληρώνει την Οδηγία 99 του 2011 που αφορά αντίστοιχα μέτρα προστασίας στον τομέα του ποινικού δικαίου. Στο τελευταίο μας Συμβούλιο ΔΕΗ στις 7 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο υιοθέτησε γενική προσέγγιση για την πρόταση αυτή και αναμένεται ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα αρχίσει τις επαφές μαζί σας για την όσο το δυνατό πιο γρήγορη υιοθέτηση της πρότασης κανονισμού. Στρέφομαι τώρα στην πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των σημαντικών εξόδων και την υπέρβαση των πολλαπλών εμποδίων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πιστωτές στη διασυνοριακή ίσπραξη των οφειλών τους. Ο προτινόμενος κανονισμός θα θεσπίσει μια νέα ενιαία και αυτοτελή ευρωπαϊκή διαδικασία για διασυνοριακές υποθέσεις, η οποία υπό ορισμένε προσεκτικά διατυπωμένες προϋποθέσεις, καθώς και με τις απαραίτητες εγγυήσεις για τον οφειλέτη, θα παρέχει στον πιστωτή την δυνατότητα να επιτύχει την έκδοση μιας ευρωπαϊκής διαταγής με την οποία θα δεσμεύει τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε άλλο κράτος μέλος. Η Κυπριακή Προεδρία πιστεύει ότι ο κανονισμός αυτός μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη επειδή θα διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή ανάκτηση οφειλών και κατ' επέκταση τις διασυνοριακές συναλλαγές. Για τον λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που σήμερα αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στον κανονισμό αυτό. Πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό αριθμό συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας και κατά τις οποίες, συμπληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση της πρότασης της Επιτροπής και προχώρησε αρκετά η δεύτερη εξέδαση του νέου κειμένου της Κυπριακής Προεδρίας. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την πρόταση αυτή τόσο στο άτυπο Συμβούλιο ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στη Λευκοσία, όσο και στο Συμβούλιο ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στο Λουξεμβούργο. Το αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών ήταν η υιοθέτηση πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών στο τελευταίο μας Συμβούλιο ΕΔΕΗ του Δεκεμβρίου. Οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν υιοθετηθεί αναφέρουν ότι ο πολιτικός στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας για την έκδοση της ευρωπαϊκής διαταγής. Περαιτέρω, ο κανονισμός θα εφαρμόζεται μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις και το στοιχείο της έκπληξης θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να διασφαλιστεί η χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Διαταγής. Τέλος, το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη όπως διασφαλιστεί ταυτόχρονα και το απαραίτητο ισοζύγιο μεταξύ των δικαιωμάτων των πιστωτών και των οφηλετών. Η υιοθέτηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών θεωρούμε ότι θα βοηθήσει την επίταξη ουσιαστικής, ουσιαστικής πρόοδου κατά τη μελλοντική εξέταση της πρότασης αυτής. Οι δύο προτάσεις κανονισμών για τις περιουσιακές διαφορές συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων αποτέλεσαν ακόμα μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Οι δύο αυτοί κανονισμοί προτάθηκαν εκ παραλίλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2011 και καλύπτουν τις διαφορές μεταξύ των πρώην συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η Κυπριακή Προεδρία έδωσε προτεραιότητα στους δύο αυτούς κανονισμούς. Προγραμμάτισε τέσσερις διήμερες συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας καθώς επίσης και ένα μονοήμερο συνέδριο στη Λευκοσία τον Οκτώβριο, στο οποίο σεμινάριο ένας από τους ομιλητές ήταν και η ραπορτέρ της Επιτροπής σας, κυρία Αλεξάνδρα Τάιν. Κατά τις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου, εξετάστηκαν εκ παραλίλου, εκ και εις βάθος και οι δύο προτάσεις κανονισμών και ολοκληρώθηκε η τρίτη ανάγνωση του αναθεωρημένου κειμένου που ετοίμασε η Κυπριακή Προεδρία. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων επιτελέστηκε σημαντική πρόοδος και επιτεύχθη σύγκληση απόψεων σε αρκετά θέματα. Στο τελευταίο μας Συμβουλίο ΔΕΗ, με τη σύμφωνο γνώμη των κρατών μελών, υιοθετήθηκαν πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και για τις δύο προτάσεις κανονισμών, οι οποίες θεωρούμε θα οδηγήσουν στην επίτευξη σημαντικής πρόοδου στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τις προτάσεις αυτές. Οι γενικές αυτές κατευθυντήριες γραμμές αφορούν μερικές από τις βάσεις δικαιοδοσίας στο θέμα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και στο θέμα της αναγνώρισης αποφάσεων προτείνει ότι θα ακολουθηθούν οι ίδιες γενικές αρχές που περιέχονται στον πρόσφατο κανονισμό για την κληρονομική διαδοχή. Επίσης, προβλέπουν ότι η ομάδα εργασίας θα εξετάσει τον βαθμό στον οποίο οι γενικές γραμμές του κανονισμού για συζύγους ακολουθούν και στον κανονισμό για τους κατοχυρωμένους συντρόφους. Η Κυπριακή Προεδρία άρχισε τη συζήτηση για την πρόταση κανονισμού για το κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων. Αν και το θέμα δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες μας, Εξετάζοντα το παράρτημα 1 τη πρόταση, όπω ήταν και η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών ΔΕΗ, η οποία λήφθηκε τον Ιούνιο. Όπω όλοι γνωρίζετε, πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέροντο και με σοβαρέ νομικέ προεκτάσει για όλου του εμπλεκόμενου. Ω Προεδρία, θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο να δώσουμε σε όλου τον απαιτούμενο χρόνο για να αξιολογήσουν τι θέσει του γενικά αλλά και ως προς τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τις ακούσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Η συζήτηση της πρότασης θεωρούμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί με την πρέπουσα λεπτομέρεια, σοβαρότητα και προσοχή. Αναφορικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και την πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα Δικαιοσύνη Επισημαίνουμε ότι το Συμβούλιο έχει πετύχει μερική γενική προσέγγιση στην πρόταση αυτή τον Ιούνιο του 2012. Η μερική γενική προσέγγιση κάλυψε όλο το κείμενο με εξαίρεση δύο ζητήματα. Πρώτο, τα ποσά του προϋπολογισμού και δεύτερο, το ερώτημα αν μερικές πτυχές της πολιτικής περί ναρκωτικών θα πρέπει να καλύπτονται από το πρόγραμμα δικαιοσύνη. Όσον αφορά τα ποσά του προπολογισμού, πραγματοποιείται διαπραγμάτευση σε οριζόντιο επίπεδο. Σχετικά με τα ναρκωτικά, η Προεδρία βρίσκεται στο διάστημα αυτό, το διάστημα αυτό σε συζητήσεις για να λύσει το πρόβλημα και είναι αποφασισμένη να εξεύρει μια λύση μέχρι το τέλος του χρόνου. Για το θέμα αυτό Κρίνοντας από τις μέχρι σήμερα επαφές με τους εισηγητές της Επιτροπής Γιούρι και Λίπε, φαίνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με το Συμβούλιο αναφορικά με πολλά κέρια ζητήματα, όπως το γεγονός ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση των δικαστών. Το Συμβούλιο, ανταποκρινόμενο και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για την κατάρτιση δικαστών έχει αναδείξει το θέμα αυτό το οποίο αποτελεί τώρα ένα από τους πιο ειδικού στόχους του προγράμματος. Αναντίλεκτα, η, κατάρτιση των δικαστών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στην προαγωγή ενός ευρωπαϊκού δικαστικού πνεύματος και δεν πρέπει να επηρεάζεται μόνο, να περιορίζεται μόνο στους δικαστές αλλά να επεκτείνεται και στους δικηγόρους, δημόσιους κατηγόρους και άλλο δικαστικό προσωπικό. Κατά την επιλογή δράσεων προς χρηματοδότηση, η Επιτροπή οφείλει να αξιολογεί τις προτάσεις με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Στα κριτήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των προτινόμενων δράσεων. Οι δίχτες έχουν αναδιατυπωθεί και διασαφινιστεί, ούτως ώστε να παρέχουν ξεκάθαρη βάση για παρακολούθηση και αξιολόγηση. Ενέκα τη εξαίρετη συνεργασίες μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και τη Κυπριακή Προεδρία, οι τριλόγοι ξεκίνησαν αμέσως μετά την ψηφοφορία προσανατολισμού στις 27 Νοεμβρίου 2012 και για του τριλόγους αυτού σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δύο τρίλογοι επί της πρότασης αυτής και έχει επέλθει συμφωνία σε σωρία ζητημάτων. Οι εργασίες για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη προχώρησαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας συμπεριλαμβανομένης και της τρίτης έκδοσης της πύλης που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 όπου προστέθηκαν νέες λειτουργίες. Ειδικότερα Όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικτυακής πύλης, προωθήθηκαν τα ακόλουθα θέματα. Πρώτον, η μεταφορά από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Δεύτερον, μια καταρχή συμφωνία για μεταφορά στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε ποινικέ υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Τρίτον, συμφωνία σχετικά με την μεταφορά της βάσης δεδομένων του Ευρωπαϊκού Αρμόδιου Δικαστηρίου από τον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα όσον αφορά αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Και τέταρτον, στρατηγική επικοινωνίας με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Μια ειδική εκστρατεία προώθησης έχει προγραμματιστεί για το 2013. Η διαδικασία προώθησης θα περιλαμβάνει μια διαφημιστική καμπάνια σε νομικά περιοδικά και άλλα σχετικά έντυπα καθώς και δραστηριότητες στρατηγικού χαρακτήρα για την προώθηση της πύλης που θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει διαφημίσεις σε κοινωνικές πλατφόρμες μέσω μαζικής ενημέρωσης και οπτικοακουστικό υλικό. Άλλες δραστηριότητες προώθησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών του 2013 είναι, είναι ακόμα υποσυζήτηση. Υπενθυμίζεται επίσης ότι μια νομοθετική πρόταση σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη αναμένεται από την Επιτροπή στις αρχές του 2013. Η πρόταση αυτή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από όλους μας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το τρέχον σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη που εγκρίθηκε το 2018 λήγει στο τέλος του 2013. Ως εκ τούτου το επόμενο έτος θα περιλαμβάνει εκτός από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημαντικές περαιτέρω εργασίες στον τομέα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης όσον αφορά το χειρισμό της νέας νομοθετικής πρότασης και την προετοιμασία ενός νέου σχεδίου δράσης για την περίοδο μετά το 2013. Το επόμενο θέμα, το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αν και το θέμα αυτό δεν είναι ανάμεσα στα θέματα που χειρίζομαι, θεωρώ ότι θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ στο έργο που επετέλεσε η Επιτροπή σας για την επίδεξη αυτής της σπουδαίας συμφωνίας. Η Προεδρία μας ευχαριστεί και πάλι τους εισηγητές του πακέτου διπλωμάτων ευρυσιτεχνίας κυρίους Λένεν, Ράπχεϊ και Παλτασάρε καθώς Χωρίς τη δική του συνδρομή δεν θα ζούσαμε αυτές τις ιστορικές στιγμές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι σήμερα οι δύο κανονισμοί υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος και παραμένει η υπογραφή τους αύριο από τους Προέδρους μας. Τώρα το μόνο που απομένει είναι η υπογραφή και η κύρωση της συμφωνίας του ενιαίου δικαστηρίου η οποία ελπίζω και εύχομαι να πραγματοποιηθεί ως έχουμε προγραμματίσει στις 18 Φεβρουαρίου 2013. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στενή και επικοδομητική συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας προς επίτευξη του κοινού στόχου της περαιτέρω εδραίωσης ενός χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας προς διευκρίνηση ουδίποτε ζητήματος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Πολύ εντυπωσιακό ο απολογισμό. Σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά για την ε, καλή συνεργασία και ιδιαίτερα αυτή την τελευταία εβδομάδα ήμασταν παρόντες με τους συγκητές και ο και συζητήσαμε τα θέματα του κανονισμού. Τώρα έχουμε αυτή τη βδομάδα τον κανονισμό για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Δύο μεγάλες επιτυχίες, πιστεύω, που οφείλονται σε εσά και που αποτελούν σημαντικά ορόσημα αυτής της πορείας. Και βλέπουμε ότι η Προεδρία που έχει το δεύτερο εξάμεινο ενός έτους ίσως δουλεύει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από εκείνη που πτυχαίνει να πέσει στο πρώτο εξάμεινο, ίσως γιατί έχει λιγότερο χρόνο στη διάθεσή της και έτσι πιέζεται και κάνει πιο πολλή δουλειά από ότι ε, θα της επέτρεπε ίσως ο πιο πολλή χρόνος. Ε, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε και πάλι και ρωτώ ποιο θέλει να λάβει για να υποβάλει ερωτήσει. Σταντέου. η κυρία Τάουν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τα όσα είπατε. Ιδιαίτερα θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός, το ότι για αυτούς τους τόσους λίγους μήνες ε, που είχαμε για τη συνεργασία με την Κυπριακή ε, Προεδρία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι διότι έπραξαν αυτά τα οποία μας είχαν υποσχεθεί, υλοποίησαν το πρόγραμμά τους και ήταν εξαιρετική η δουλειά και η συνεργασία. Και ιδιαίτερα για τα δύο αυτά μεγάλα νομοθετήματα νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πολύ περήφανοι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και εύχομαι κάθε επιτυχία και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τσέον. Ναι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ θερμά την Κυπριακή Προεδρία. Τα δύο θέματα που με ενδιαφέρουν εμένα, ε, το, δικαίω, το δίκαιο το σχετικό με τα αγαθά, έχουν προχωρήσει πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυπριακή Προεδρία για, την, ε, για το ενδιαφέρον που έδειξε και η διάσκεψη στη Λευκοσία μας βοήθησε να προχωρήσουμε πολύ, ήταν πολύ σημαντική και για μένα. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω ότι ιδιαίτερα η ε, αποκάλυψη για μένα ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η επιλογή των προσώπων για τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να προχωρήσει καλά και αποτελεσματικά. Και άλλα θέματα προχωρήσανε παρότι ήταν πολύ περίπλοκα. Πρέπει να σας πω ότι επειδή και μικρό κράτος είστε δεν περίμενα τόσα πολλά από την Κυπριακή Προεδρία, αλλά πάντως στα θέματα που εμένα με αφορούν είχατε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βίξτρο. Σας ευχαριστώ θα ήθελα και εγώ να εκφράσω ειλικρινή, ειλικρινείς ευχαριστίες. Ξέρουμε ότι η Κύπρος είναι μια όμορφη χώρα, ένα, μικρό, ένα όμορφο νησί, μικρό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά αυτή η εικόνα νομίζω ότι αρχίζει και οχριά σιγά σιγά, καθώς βλέπουμε ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει αφήσει την εντύπωση ότι είναι όχι απλώς μια μικρή όμορφη χώρα η Κύπρος, αλλά πάνω απ' όλα μια πολύ σημαντική χώρα για την Ευρώπη διότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας αυτής κάνατε ρηξικέλευθο έργο. Ανοίξατε παιδεία καινούρια όπως ε, το θέμα παραδείγματι της ευρεσιτεχνίας που είχε χρονίσει και μπορέσατε εσείς να το ολοκληρώσετε με μεγάλη επιτυχία ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα μας πάει θα μας υποχρεώσει σε μερικές δεκαετίες ακόμη να θυμόμαστε εκείνε τι μέρες της Κυπριακής Προεδρίας και να λέμε να, μια μικρή χώρα που είχε τόσο σημαντική, τόσο ζωτική σημασία για την Ευρώπη. Ιδιαίτερα για τόσο σημαντικά θέματα και μπορούμε νομίζω να το πούμε αυτό τώρα που κλείνει και η Κυπριακή Προεδρία, η περίοδος της Προεδρίας σας, άλλα θέματα όπως το πακέτο για το άσυλο, το οποίο επίσης πιστεύουμε ότι μπορούμε να δούμε να ολοκληρώνεται σιγά σιγά πάλι έχει αφήσει το στίγμα της η Κυπριακή Προεδρία. Όπως είπα και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε την Κύπρο στο μυαλό μας σε μια πολύ σημαντική για την Ευρώπη χώρα. Σας εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες και εύχομαι τώρα πολύ καλή ανάπαυση ύστερα από την τόση σκληρή δουλειά που κάνατε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, ε, δεν ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε. Συνήθως κύριε Πρόεδρε απολογούμαστε γιατί, για το τι δεν έχουμε κάνει. Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος και ευχαριστημένος γιατί καταφέραμε τουλάχιστον αυτά που είχαμε υποσχεθεί να τα εκπληρώσουμε. Είμαστε μικρή χώρα, εκτός από αυτά που έχουμε κάνει ελπίζω να σας να καταλάβετε και την κυπριακή φιλοξενία όσοι επισκεφθήκατε την Κύπρο και ε, ο σκοπός μας είναι κοινό. Η Ευρώπη ένας χώρος ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ κύριε Υπουργέ. Ήταν πολύ όμορφη η συζήτηση και εύχομαι και καλές γιορτές τώρα πλέον και πολύ καλή χρονιά. Και προχωρώ με το υπόλοιπο της ημερησίας διατάξεως, γιατί κανονικά... Α, όχι, τώρα έχουμε την έκθεση της κυρίας Ρότσπεραντς, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όταν ορίστηκα συγκέντρια εκ μέρου τη Επιτροπή μα για το θέμα των, ε, του δημοσιοπαλληλικού κώδικα και του κανονισμού μάλλον υπηρεσιακή κατάσταση, θεώρησα ότι το θέμα αυτό θα είχε κλείσει λίγο πολύ και ότι ίσως θα ήταν ε, σκόπιμο να προβλέψουμε απλώς μια μικρή επισκόπηση προς το τέλος της χρονιάς για να σας πω πού βρισκόμαστε. Και θα ήλπιζα, θα ήλπιζα να μπορούσα να σας αναφέρω κάτι το πραγματικά καινούριο, κάτι το νέο. Στην τελευταία συνεδρίασή μας ε, με τους κοιόδης συγκητές στο Στρασβούργο, Πρέπει να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεδρίαση, συναδελφικό πνεύμα και όλα αυτά. Αλλά πρέπει να πω ότι οι συνάδελφοι πάντα ρωτάνε Ωραία, τι καινούριο έχει να μα πει. Ε, Δυστυχώ λοιπόν δεν έχω τίποτα νέο να σα πω. Κάτι καινούριο όμω από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι σήμερα ε, υπάρχει τουλάχιστον εκ μέρους του Συμβουλίου μπορώ να πω σας δύο λόγια μόνο ουσιαστικές αλλαγές από πλευράς του Συμβουλίου στις επίσημες επαφές με κάποια προεδρία δεν υπάρχουν τριμερής διάλογος δεν έχει λάβει χώρα η Κυπριακή Προεδρία δεν έλαβε διαπραγματευτική εντολή για τα κράτη-μέλη περιμένανε μια απόφαση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ελπίζαμε ότι 22 και 23 Νοεμβρίου θα μπορούσε να ληφθεί μια απόφαση έτσι ώστε να διευκρινιστεί κάπως η κατάσταση και να δούμε τι είδους περιθώριο χειρισμών έχουμε και για άλλα ζητήματα. Πλην όμως, τώρα κοιτάμε περισσότερο για τις 6 και 7 Φεβρουαρίου το επόμενο ραντεβού. Πάντω πρέπει να πω ότι η Κυπριακή Προεδρία και προ το τέλο ακόμη της θητεία της και σήμερα έχει καταθέσει ε, για το Κορεπέρ μια έκθεση προόδου. Μια έκθεση προόδου η οποία περιλαμβάνει λίγες αλλαγές σε σχέση με την έκθεση πρόοδου της Προεδρίας της Δανίας, η οποία επίσης είχε, όπως ξέρετε, το θέμα αυτό. Κάποια μικρά ζητήματα που είχαν ήδη κάπω ε, σχεδιάσει οι Δανείοι, αλλά για τα οποία ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί πλειοψηφίε ή σαφήνεια. Για τους συμβασιούχου, για παράδειγμα, contract agents, όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει. Μια τη μέθοδο, method, το ζήτημα πάνω απ' όλα του ποιο είναι το μέγιστο του υπολογισμού της μεθόδου προσαρμογής. Υπάρχουν κάποιες ιδέες. Στην έκθεση πάντως προόδου ε, υπάρχει κάτι το πολύ ωραίο και θα θέλω να σα διαβάσω και στο αρχικό του κείμενο, γιατί αναφέρεται στις συντάξει με προτινόμενη ηλικία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω λέει η Προεδρία, το κείμενο αυτό τη Προεδρία, ότι είναι εντάξει. Αλλά σα διαβάσω τώρα στα αγγλικά. Συνεχίζουν. Πλην όμω, συσχετισμό μεταξύ τη ηλικία συνταξιοδότηση και. Ε, προσδόκιμου ζωή θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Ενώ θα πρέπει να καταργηθεί η πρόορη ταξιοδότηση χωρίς, ε, ε, ε, επιβάρυνση. Προφανώ υπάρχουν κράτη τα οποία θέλουν να συσχετήσουν την ηλικία τη συνταξιοδότηση με το προσδόκιμο ζωή. Πολύ φάνταστο μου φαίνεται αυτό, αλλά εν πάση υπάρχουν κράτη τα οποία ζητούν όλο και περισσότερα για περικοπέ στο προσωπικό προβλέπεται το 5% από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα αναφέρεται στις προτάσεις εδώ στην έκθεση πρόοδο ότι να το ελάχιστο αυτό το 5%. Μετά έχουμε 20 Δεκεμβρίου, μεθαύριο ουσιαστικά, τη συζήτηση και πάλι στο ε, Συμβούλιο. Πάντως η έκθεση προόδου μόνο ε, παρελήφθη από το Κορεπέρ, λήφθη, ε, έλαβε γνώση το Κορεπέρ, καταγράφει την κατάσταση μόνο τίποτε περισσότερο και δεν έχει δοθεί, όπως είπα, ούτε ακόμη και μετά την έκθεση αυτή, εντολή διαπραγμάτευσης, παρότι έχουν παρέλθει 8 μήνες. Ε, τον Φεβρουάριο, όπως είπα, συνεδριάζει το Συμβούλιο. 11 Φεβρουαρίου ομάδα εργασίας της Ιρλανδικής πλέον Προεδρίας και εξαιτίας των αποτελεσμάτων της, ε, προεδρίας της συνεδρίασης του Συμβουλίου θα προβλεφθούν ταχύτατα, ελπίζω, ε, συνεδριάσεις του τριμερούς διαλόγου. Τα ζητήματα τα γνωρίζουμε βέβαια όλοι. Ε, έχει εδώ και καιρό καταστεί σαφές ότι ένα μέρος του κανονισμού δημοσιοϊπαλληλικής κατάστασης ε, που αφορά τη μέθοδο και την προσαρμογή των, τη μέθοδο προσαρμογής των ε, μισθών και ιδιαίτερα τον το ειδικό τέλος special levy ονομάζεται για την αντιμετώπιση της κρίσης ξέρουμε ότι πνέων στις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου δεν υπάρχει πλέον μέθοδος προσαρμογής για το 2013 εφόσον δεν υπάρχει νέα νομοθεσία και επίσης από 1η Πρώτου του 2013 δεν υπάρχει αυτή η εισφορά αλληλεγγύης. Ο κύριος Σεύκοβιτς, ο αρμόδιος επίτροπος, στις 30 Νοεμβρίου, απευθυνόμενος ε, με επιστολή στον πρόεδρο Σούλτσο και την Κυπριακή Προεδρία, τον κύριο Μαυρογιάννη, καλεί το Συμβούλιο και το Κορεπέρ να χορηγήσουν παράταση της ισχύω της μεθόδου προσαρμογή και του ειδικού τέλους ε, ε, κατά ένα, έτος ακόμη μέχρι ότεθεί σε ισχύ ο νέος κώδικας δημοσιοπολιτικής κατάστασης έτσι ώστε τον Ιανουάριο να μην αντιμετωπίσει το ζήτημα της αυτόματης αναπροσαρμογής προς τα άνω των ε, μισθών δεδομένου ότι δεν θα είναι πλέον νόμιμη η παρακράτηση του τέλους αλληλεγγύης ή της εισφοράς αλληλεγγύης καλύτερα. Το Κορεπέρ στην συνεδρίαση την προπροηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη-τελευταία εβδομάδα, την ε, πέμπτη δηλαδή πριν από το Στρασβούργο, συνεδρίασε και με μια, σε μια συνεδρίαση που καθένας την περιγράφει διαφορετικά, ανάλογα με το με ποιον μιλάτε, από το πρωινό μέχρι το βραδινό άλλες ε, εντυπώσεις περιγράφονται, κατέληξε ότι μπορεί να παραταθεί μεν η εισφορά αλληλεγγύης, αλλά όχι η μέθοδος αναπροσαρμογής των νηστών Εδώ μιλάμε για, παιδι... για νηπιαγωγείο, εδώ μιλάμε για νοησίες. Μέχρι τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, τόσο ή άλλως θα υπάρχει ε, νέα νομοθεσία και θα αρχίσει πάλι να υπολογίζεται από τον Ιούλιο το αργότερο η μέθοδος και να αναπροσαρμόζεται. Εν πάση περιπτώσει είναι τέτοιο νηπιαγωγείο και τέτοιο, τέτοια νοριμότητα που επιδεικνύεται που δυστυχώς όμως πρέπει να σας αναφέρω που πραγματικά δεν ξέρω αν χρειάζεται να τη συζητάμε. Μετά έχουμε την κατάσταση κατά την οποία τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ε, ειδική πλειοψηφία, μόνο για την παράταση της μεθόδου και της εισφοράς αλληλεγγύης που, δεν, ε, που ουσιαστικά αυτό που θέλανε με την ε, πρόταση ήταν να μην παραταθεί να μην αυξηθεί μάλλον αυτόματο ο μισθό. Ε, το Βέλιο και το Λουξεμβούργο βέβαια ήταν κατά, το ε, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι θέλανε να επιβληθεί αυτή η παράταση. Από αυτό που <laughs> όπως θα λέγανε οι δημοσιογράφοι μπορώ να σας πω ότι από καλά πληροφορημένες πηγές γιατί το και όχι μόνο από το Κορεπέρα αλλά και παλού υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία θεωρούν ότι δεν τους κάνει και τόσο κακό η δημοσιότητα, η αρνητική που παίρνουν οι υπάλληλοι, οι ευρωυπάλληλοι, ότι δηλαδή θα αυξηθούν αυτόματα οι μισθοί τους κατά 5,5%. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό συμφωνήσανε. Η πρόταση επιτροπή που ούτως ή άλλως ήταν πολύ περίπλοκη και εμεί βέβαια από πλευρά μα έπρεπε αμέσω να ξεκινήσουμε να διαπραγματευόμαστε πολύ γρήγορα, με τριμερή διάλογο κτλ. Ενώ εμεί είμαστε στον, στο Στρασβούργο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε οργανωθεί και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, να ανταποκριθούμε. Αλλά όπω είπα δεν εξασφαλίστηκε ε, πλειοψηφία και έτσι τουλάχιστον η Επιτροπή ακολουθώντας ε, τους κανόνες και τους κανονισμούς και τις διατάξεις ε, μιλάει για προσαρμογή των μισθών και συντάξεων είναι υποχρεωμένη λόγω της νομοθεσίας να το πράξει από 1η Ιανουαρίου. Σε αυτό πάλι δεν εξασφαλίστηκε ε, ειδική πλειοψηφία για την παράταση μεθόδου. Παρά του Λουξεμβούργου και του Βελγίου δεν υπήρχαν κράτη-μέλη που να συμφωνούσαν σε μια λύση, ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση. 118, 6-7 δηλαδή, μεγάλα και μεσαία κράτη που απήχαν της ε, και έτσι δεν εξασφαλίστηκε η δική πλειοψηφία. Τόσο λοιπόν ως εισηγήτρια αλλά και προσωπικός ετοίμασε ένα ανακοινωθέν και για τα δύο αυτά θέματα και ιδιαίτερα το ζήτημα το ότι δεν, είμαστε σε θέση, ότι δεν ήταν σε θέση το Κορεπέρ να παρατείνει την ε, αλληλεγγύη, το, την εισφορά αλληλεγγύης και άρα θα σταματήσει. Έκανα το ανακοινοθέν... ως εισηγήτρια όπως είπα επικρίνοντας την ανικανότητα των κρατών μελών, την αδυναμία τους να δούνε τα σημαντικά και την ε, αποτυχία ουσιαστικά του Συμβουλίου να προχωρήσει σε σχέση με την αιτήση αυτή προσαρμογή και αντίστοιχα βέβαια και του στεξιωτικού ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των μισθών όπως και των συντάξεων να ακολουθήσει τα όσα ορίζει η νομοθεσία. Και προβαίνω σε μια ανακοίνωση τύπου τώρα μαζί με τον συνάδελφο κ. Μπαλταζάρε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς είναι προφανές ότι απέτυχε το Συμβούλιο και πάνω απ' όλα δεν αναγνωρίζει αυτά που ορίζουν οι νόμοι, οι συνθήκες, η νομοθεσία μας. Αντίστοιχα θα κληθεί βέβαια το δικαστήριο να λάβει απόφαση. Φαντάζομαι θα γίνει προσφυγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ελπίζω ότι μεταξύ των κρατών μελών θα υπήρχαν ε, περισσότερα, τουλάχιστον σε επίπεδο πρωτευουσών, ίσω ακόμη να παραμένουν πιστά στην νομοθεσία και τι ε, συνθήκε. Αλλά φαίνεται ότι με το που παίρνουν το αεροπλάνο και έρχονται στι Βρυξέλλε, γυρνάνε το, το, παλτό μέσα έξω και αλλάζουν βιολί και μιλάνε με διαφορετική γλώσσα. Αυτή είναι η κατάσταση κύριε Πρόεδρε. Δημερό σα έχω ενημερώσει του άλλου, κύριε Πρόεδρε, όπω και του ε, σκιώδης ηγητέ. Η γραμματεία βέβαια είναι πάντα ενήμερη. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής που είναι εδώ γενικός, αναπληρωτής γενικός διευθυντής και το επιτελείο γενικά της Επιτροπής είναι εδώ παρόντες και γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Αυτή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Λίχτενμπέργκερ. Καταρχάς, συμφωνώ απολύτως με τη συνάδελφα κυρία Ρότσπεραντ για την κατάσταση όπως την περιγράφει σε επίπεδο συμβουλίου. Εγώ καταλήγω ότι αργά αργά πλέον αλλά αναπόφευκτα γίνεται αυτή η κατάσταση ανυπόφορη από πλευράς του Συμβουλίου. Βλέπουμε ότι απορρίπτει προτάσεις του, του Κοινοβουλίου ακόμα και εις βάρος των ιδίων του συμφερόντων και λησμονεί ότι όλοι μέσα στην Ευρώπη ζούμε. Δεν υπάρχουν οι κακοί στις Βρυξέλλες και οι καλοί στο Βερολίνο, τη Βιέννη, το Παρίσι και τη Ρώμη. Αυτό το λησμονεί το Συμβούλιο. Η δυσκολία που είχαμε σε όλη αυτή την ιστορία ήταν ότι λίγοι είναι αυτοί στην Ευρώπη οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν ποιο είναι το πλέγμα το θεσμικό και ποιος είναι αρμόδιος γιατί πάντα παρουσιάζεται η κακή Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι άλλωστε και το πρόβλημά μου ως προς το επικοινωνιακό κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας. Και πρέπει να πω ότι με δυσκολεύει ιδιαίτερα το γεγονό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Το έχουμε αντιμετωπίσει σε πολλά ζητήματα, σε πολλού φακέλου ε, προ διαπραγμάτευση. Εδώ όμω είναι ιδιαίτερα ε, προφανές και συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται από πλευρά του Συμβουλίου. Εμείς πάντως έχουμε συμφωνήσει, έχουμε προσδιορίσει τη θέση μας. Εκ μέρους της ομάδας μου είχα κάνει και πιο ακραίες προτάσεις. ώστε να είναι ο, το τέλος αλληλεγγύη σε πραδείγματι προοδευτικό ή να μιλήσουμε για τις, αν και δεν ξέρω αν αυτό νομικά τουλάχιστον στέκει, είναι εύκολο να, επιβληθεί, να επιβάλλουμε στις πιο υψηλές συντάξεις ενδεχομένως ένα είδος τέλους αλληλεγγύη, αλληλεγγύης και όλο αυτό το ζήτημα της αντιπαράθεσης ε, της σχετικής με το τέλος εκπατρισμού θα μπορούσαμε ενδεχομένως να το αντιμετωπίσουμε χάρη σε συγκεκριμένα ε, ποσά και όταν πια έχει περάσει πάρα πολύ χρόνος και κάποιος ε, για πολύ μεγάλο διάστημα πια ζει και εργάζεται στι Βρυξέλλες και δεν είναι σε θέση να αιτιολογήσει την ίσπραξη ε, αυτού του, αυτού του ποσού εκπατρισμού ίσως να το καταργήσουμε αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν διάφορες ιδέες τις έχουμε συζητήσει Έχουμε μια κοινή θέση εμείς από πλευρά μας Κοινοβουλίου. Αυτό που με ενοχλεί εμένα πάνω απ' όλα όμως είναι η θέση, η συμπεριφορά του Συμβουλίου, η οποία είναι επιβλαβής εν τέλει. Είναι επιζήμια και εμάς μας δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα, γιατί βεβαίως εγώ δεν, δεν βρίσκομαι σε καμιά πρωτεύουσα κράτους που να έχω όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θέση μου και να εξηγώ τις θέσεις μου ή να κατηγορώ κάποιον άλλον για τα όσα συμβαίνουν. Μπορεί σε, κάποιους άλλους, σε κάποια άλλα ζητήματα να, μπορούσε να, να, το είχαμε ήδη εντοπίσει, αλλά εδώ πια είναι καταφανή η συμπεριφορά του Συμφούλου. Ευχαριστώ, κυρία Τσάιν. Θα συμφωνήσω και εγώ, κύριε Λιχτενμπέργκερ, με τα όσα είπατε, ειδικά για το ζήτημα της... Ε, του εκπατρισμού, του ποσοστού ε, του μισθού για τον εκπατρισμό για όσους ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Βέλγιο δεν νομίζω ότι πια έχει νόημα. Άλλο θέμα τώρα για την ηλικία σταξιοδότησης ή ε, και το συσχετισμό με το προσδόκιμο ζωής. Ξέρω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε προσπαθήσει να γκρίνουμε μία έκθεση σε σχέση με ένα ενιαίο, ε, μια ενιαία ηλικία σταξιοδότησης, η οποία ακριβώς αυτό είχε αποτύχει, γιατί είπαμε μία υπουργό η οποία είχε πει ότι αν ορίσουμε ως έτος τα τα 67 έτη, τότε ε, ε, ίσως για ορισμένα κράτη, όπως το δικό μου μου είχε πει αυτή η υπουργό, ε, δεν υπάρχει λόγος καν να υπολογίσω να δώσω σύνταξη, γιατί τα 67 έτη ηλικία είναι το μέσο έτος, η μέση διάρκεια ζωής. Σλοβακία νομίζω, δεν πάει περιπτώσει κάποιο κράτο από την Ανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, όντω το είχα ψάξει τότε, είχα ψάξει και ήταν όντω έτσι. Ε, ε, από την άλλη πλευρά, εμεί στη Γερμανία φέτο την Άνοιξη μπορέσαμε να φτάσουμε στο επίπεδο που ένα πρώην ε, υπήκο τη Λαϊκής Δημοκρατίας Γερμανίας, Ανατολικής Γερμανίας δηλαδή, έφτασε τώρα 23 χρόνια μετά την επανένωση να έχει το ίδιο προσδόκιμο ζωής με τον κάτοικο των δυτικών κρατηδίων. Κάτι το οποίο μας δείχνει πόσο σημαντική είναι και η υποστήριξη των δυτικών κρατηδίων για την Ανατολική Ευρώπη. Χωρίς αυτή δεν θα είχε μπορέσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο ε, προσαρμογή στο επίπεδο ζωής ή προσαρμογή στο προσδόκιμο ζωής επίσης δεν θα έχει εξασφαλιστεί και γι' αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό δεν έχει κανένα νόημα να ζητούμε από τους ανθρώπους να κάτσουν μέχρι μια προχωρημένη ηλικία πριν πάρουν τη σύνταξη εάν πια είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν κάτι άλλο Μία πρόταση η οποία είχε απορριφθεί, αλλά είχα υποβάλει εγώ την ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να, υποβληθεί να, να συμπληρωθεί μάλλον ε, το προσωπικό με μια επιπλέον κατηγορία που θα ήταν γραμματιακή. Ε, το θέμα αυτό έχει παραμείνει στις συζητήσεις ή το έχουν απορρίψει και έχει φύγει τελείως από την τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος. Ναι, να, ζητήσω, να πω και εγώ δύο λόγια γιατί Πιστεύω ότι πρέπει να υποθούν ορισμένα πράγματα πολύ ξεκάθαρα. Αυτή η αύξηση του 5,5% που θα γίνει αναγκαστικά θα γίνει ευθύνη και μόνο του Συμβουλίου, εκείνων των κρατών δηλαδή τα οποία απέσυραν την υποστήριξή τους ως προς την πρόταση του Επιτρόπου ε, Σεύκοβιτς. Αυτό το 5,5% δεν έχει σημασία αν είναι αύξηση ναι ή όχι, ε, εάν είναι ουσιαστική πραγματική αύξηση ή όχι. Το μόνο σημαντικό είναι ότι δίνει την ευκαιρία στον κίτρινο τύπο να αναπτύξει μια νέα πολεμική, μια νέα σειρά επιθέσεων εις βάρος των ευρωϊπαλλήλων. Ε, επίσης πρέπει να περιμένουμε πολύ σύντομα και την επόμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του σχετική με την μέθοδο προσαρμογής, όπου πάλι θα αποφασίσει το ίδιο πράγμα που είχε αποφασίσει και την προηγούμενη φορά το δικαστήριο και φαντάζομαι και τρίτη φορά στην ίδια αποφάση θα καταλήξει, γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με απλή καταστρατήγηση του δικαίου. Τίποτε άλλο παρά καταστρατήγηση του δικαίου. Πράγμα το οποίο θα ήταν ποινικά κολάσιμο στη δική μου την ε, πατρίδα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορεί δηλαδή κανεί να περιμένει ότι τα κράτη-μέλη προχωρούν ε, σε ένα ζήτημα το οποίο έχει κρυφθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και παραβιάζοντας την ε, δικαιοσύνη, την νομοθεσία αγνοούν την απόφαση του δικαστηρίου, αγνοούν τους ισχύοντες κανόνες και δεν την εφαρμόζουν. Έτσι λοιπόν, όταν έχει αποφασίσει ομόφωνα το Συμβούλιο, γιατί κάθισαν όλοι και συζήτησαν και έγνευσαν καταφατικά και είπαν ναι, ναι, αυτό θα κάνουμε. Ε, μάλλον τώρα λοιπόν θα βρεθεί ο τρόπος να προβληθεί αυτό μέσω των μέσων μαζική ενημέρωση κατά πολύ ε, στρεβλό τρόπο. Ένα δε από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε, και αυτό το αναφέρω και αυτό και το οποίο το έχω δει και από διάφορε συζητήσει όλους αυτούς τους μήνες, σε κράτη-μέλη και στην δική μου την πατρίδα βέβαια. Μεγάλο μέρος του προβλήματος λοιπόν έχει να κάνει με ένα, μια απλή παιδιαρίστικη ζήλια ορισμένων δημοσίων υπαλλήλων των κρατικών υπηρεσιών των ε, κρατών αυτών, των κρατών μελών, ει βάρο των ευρωϋπαλλήλων. Κάθονται στα γραφιάκια του δηλαδή και λένε Α, αυτοί εκεί πέρα χρυσοπληρωμένοι κτλ. Και, και έτσι φτιάχνουν όλο αυτό το πλέγμα, όλο αυτό το πνεύμα. Ένα πλέγμα και ένα πνεύμα που προφανώ δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί και το οποίο οδηγεί σε προβλήματα έστω κι αν ε, σε ορισμένε περιπτώσει έχει μπορέσει η μέθοδο σε παραδείγμα, να, κάνει, να οδηγήσει σε μια προσαρμογή ε, των μισθών. Αυτό είναι το πρόβλημα πάνω απ' όλα που αντιμετωπίζουμε. Τώρα, έχουμε επίση την εκκρεμότητα αυτή των έξι μηνών. Εμεί έχουμε προσδιορίσει τις θέσεις μα, Έχουμε δώσει την αντολή για τη διαπραγματεύση πρώτη ανάγνωση. Δεν έχει προχωρήσει η κατάσταση διότι παρεμποδίζει το Συμβούλιο. Η κυρία Ροτ ε, Πέρεντ ασφαλώ θα απαντήσει τώρα την ερώτηση τη κυρία Στάιν, αλλά εγώ θα επισημάνω δεν γίνεται τίποτα γιατί δεν συζητεί σοβαρά το Συμβούλιο. Ούτε καν τάσει δεν διαβλέπονται για, να, για διαμόρφωση μια κοινή θέση, μια πλειοψηφία, μια συγκεκριμένη εντολέ. Όλα ε, εντοπίζονται στο ζήτημα του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά ερωτώ εγώ ποιο θεωρεί ότι μπορεί να, ε, να υποαγορεύσει με όμοιρο το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο το κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. Όποιο το έχει φανταστεί αυτό, απατάτε πλάνιν ικτράν και εγώ σας βεβαιώ ότι θα μπορέσουμε να επιδείξουμε, να αποδείξουμε πόσο τα λεγόμενα αυτά προνόμια είναι ε, σωστά, είναι απαραίτητα και δεν θα αφήσουμε να παρασυρθεί όλη αυτή η κατάσταση σε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό δημο, ε, δημόσιας διοίκησης ο οποίος θα λειτουργεί ικανοποιητικά που θα λειτουργεί σωστά. Αυτές ήταν οι δικές μου σύντομες παρατηρήσεις. Κυρία Συγγήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ολόψυχα, wholeheartedly και απόλυτα μπορώ να υπογραμμίσω και εγώ τα όσα είπατε γιατί πρέπει να πω ότι μου φαίνεται αδιανόητο το να υπάρχει νομοθεσία, κανονισμός υπαλληλική καταστάσεως με τη μέθοδο προσαρμογής, με τους λοιπούς κανονισμούς και διατάξεις που ισχύουν και που ομόφωνα όπως και εσεί επισημάνατε τώρα ε, εγκρίθηκε την περίοδο 2003-2004, τέθησε εφαρμογή το Μάιο του 2004 συγκεκριμένα και Τώρα τα κράτη συμπεριφέρονται σαν να μην έχουν καμία ανάμειξη σε όλη αυτή την υπόθεση. Τα παλαιά κράτη-μέλη την έχουν λησμονήσει, τα δε νέα συμπεριφέρονται σαν να μην ισχύει για αυτά το κοινοτικό κεκτημένο, σαν να φτιάχνουμε μια Ευρώπη à la carte και ο καθένα να παραγγέλνει όποιο κομμάτι τον βολεύει. Και αναλόγω και οι προσαρμογέ των μισθών δείχνουν ότι πρέπει βεβαίω να γίνει ε, ο υπολογισμό με βάση τη μέθοδο. Για να δούμε λοιπόν ε, την κατάσταση σε σχέση με τα κράτη-μέλη, τα λεγόμενα ε, του καλαφιού, δηλαδή τα βασικά κράτη-μέλη, τα οποία έχουν για το 2012 4,3 αύξηση 4,3 η Γερμανία, 4,5 το Βέλγιο, 2,5 το Λουξεμβούργο, 1,8 η, η Γαλλία στους ε, ε, μισθούς. Ενώ η Βρετανία έχει μόνο 0,9 αύξηση, 0,9%, ε, μηδενική αύξηση η Ιταλία, μείωση 1,9% ε, οι κάτω χώρε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η βασική ιδέα. Εδώ πέρα συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε, με εσά ότι το πρόβλημα πάνω απ' όλα εντοπίζεται σε αυτά τα ε, αισθήματα ζηλοτυπία ορισμένων κρατικών δημοσίων υπαλλήλων. Για το κομμάτι του σχετικό με τις εξοικονομήσεις δεν έχω τίποτα να, να σχολιάσω. Για δε τις ε, συντάξεις θα ήθελα να πω ότι δεν θεωρώ ότι μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με το προσδόκιμο ζωής θα μπορούσε να φτάσει κανείς στο σημείο κάθε χρόνο να κοιτάει τα στατιστικά στοιχεία, να βλέπει ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής και αναλόγως να προσαρμόσει για ένα-δύο χρόνια την ηλικία ταξιοδότηση. Αυτό οποιοδήποτε νομικό θα μα πει ότι δεν στέκει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητούνται ανα πάσα στιγμή τα, ε, οι απαιτήσει και οι προσδοκίε ε, ενό εργαζομένου. Για να δούμε τώρα το επίδομα εκπατρισμού, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Για να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό μπορεί για τον καθένα να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Αλλά το να σκεφτούμε ότι με το να δουλέψει κανείς για 10 χρόνια σε μια θέση εργασίας. Σημειώνω δε ότι πριν δεν μπορεί να έχει ζήσει στο Βέλιο, διαφορετικά δεν θα δικαιούται το επίδομα εκπατρισμού. Δηλαδή ήρθε τα τελευταία 10 χρόνια στις Βρυξέλλες και βέβαια πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερως ότι εξετάζεται με πολύ μεγάλη αυστηρότητα που ήταν εγκατεστημένος πριν που δούλευε. Και άρα έρχεται και παίρνει αυτό το επίδομα εκπατρισμού για το οποίο θα ήθελα να λάβετε υπόψη τα εξής δύο στοιχεία. Η μέση η ηλικία ανάληψης ε, της θέσης είναι 25-35 έτη. Έτσι. Άρα μέσα στα 10 χρόνια τι έχουμε υπαλλήλους 35 με 45%. Και εκείνη την ώρα τους κόβεται κατά 16% το εισόδημα. Τι περιμένετε ότι θα κάνουν. Θα έχουν όλη αυτή την εμπειρία συσσωρεύσει επί 10 χρόνια. Ε, οι πιο καλοί θα σηκωθούν να φύγουν και θα πάνε αλλού. Θα πάνε σε εταιρείε παροχή συμβουλών, σε consulting, στη βιομηχανία κτλ. Θα χάσετε δηλαδή τους πιο ικανούς, τους πιο, τους πιο Οι λιγότερο ικανοί δεν έχουν άλλη επιλογή και μένουν στα θεσμικά όργανα. Αυτό θέλουμε. Πρώτο το ερώτημα. Δεύτερο, και να μιλήσουμε για τι διπλωματικέ υπηρεσίε. Οι διπλωματικέ υπηρεσίε βεβαίω έχουν υψηλό επίδομα εκπατρισμού και όχι επειδή περνάνε πότε πέντε χρόνια στην Αφρική, πότε τρία χρόνια στο Βέλγιο και πότε επτά χρόνια στο Μεξικό. Το παίρνουν, παίρνουν και την ε, ε, φοροαπαλλαγή για τις ε, αγορές τους, όλα αυτά τα προνόμια τα οποία προσπάθησε το Κορεπέρ να μας αποκρύψει και από εμάς και από τον Πρόεδρο κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουμε παρά σε όλα αυτά δεν έχουμε παρά να δώσουμε την εξή απάντηση. Να κόψουν αντίστοιχα τις, ε, τα, τα επιδόματα εκπατρισμού από τι διπλωματικέ του υπηρεσίε, τα κράτη-μέλη. Το να λέμε ότι δεν το κάνουμε για την ε, μόνιμη αντιπροσωπεία. Το να λέμε ότι δεν το κάνουμε για τι εθνικέ δημοσ... ε, διπλωματικές υπηρεσίες. Αλλά το κάνουμε για τους ευρωϊπαλλήλους. Τότε μόνο για σύμπλαγμα μπορώ να μιλάω. Για σύμπλαγμα κατητερότητα και για ζήλια. Εγώ αυτό που θέλω είναι να έχω τους καλύτερους υπαλλήλους, το καλύτερο προσωπικό στη διαδεσή μου. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι δυνατόν να το εξασφαλίσω αυτό και να απαιτώ, γιατί ξέρω όταν έχω κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει, έχει μάθει τη δουλειά καλά, είναι κρίμα να τον χάνω και γι' αυτό εγώ δεν θέλω επουδενή να καταργηθεί αυτό το επίδομα εκπατρισμού. Είμαι διατεθειμένη μέχρι τέλος να το υποστηρίξω. Για, το... για την εισφορά αλληλεγγύης. Και έχει δίκιο ο κύριο Προεδρό, ότι τα κράτη-μέλη αυτή την ε, περίοδο την ε, έχουν ε, ε, ούτως ή άλλως την, έχουν γραμμένη στα παιδιά του στα παπούτσια αυτή την εισφορά ε, αλληλεγγύη, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι μέσα σε τρει-τέσσερι μήνες, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος πολύ σωστά, θα επανέλθει. Επομένως αυτού του τρει-τέσσερι μήνες κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αξιοποιούν δηλαδή αυτή την ιδέα, το χρησιμοποιούν ως εργαλείο, ως μέσον για να ε, κυκλοφορήσουν δυσμενείς ειδήσει και να αμαυρώσουν ε, την εικόνα του Κοινοβουλίου και των υπαλλήλων γενικότερα. Βέβαια αυτό χρειάζεται πολύ γερά νεύρα. Νεύρα γερά έχω εγώ, επιμονή και υπομονή έχω, δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Θα εμείνω και θα είμαι πάντα στους αγώνες. Το θέμα τώρα είναι αν μπορεί αυτό, αυτή η σφορά αλληλεγγύης να αλλάξει. Βεβαίως και μπορεί να αλλάξει. Βεβαίως. Μπορεί να την πάμε μέχρι το βαθμό 16 μέχρι το 16ο βαθμό. Να το δεχθώ, να το συζητήσω. Αλλά για να το λάβω, για να το κάνω αυτό, τότε θέλω και κάποιο αντάλλαγμα. Χωρί αντάλλαγμα δεν γίνεται. Και πρέπει πάλι απ' όλα να πω, και ζητώ συγγνώμη, Εύα, ε, αυτό που δεν δέχομαι είναι να περικοπούν de facto οι συντάξει. Κάποια στιγμή ίσω να μα πει η Επιτροπή ποια είναι τα στοιχεία θα έπρεπε εγώ να τα γνωρίζω τα στοιχεία, ομολογώ, αλλά ε, δεν τα έχω πρόχειρα. Λοιπόν, να μας πει ποια είναι τα ποσοστά, τα μέγιστα ποσοστά ε, συνταξιοδότησης. Αυτοί που φεύγουν, που φεύγουν κάπου σε, σε μια μέση βαθμίδα ε, του management και δεν ξεπερνούν και το 70% ως ποσοστό επί του μισθού για τη σύνταξη. Ε, λοιπόν, δεν νομίζω ότι σε αυτούς μπορούμε να κάνουμε περικοπές σύνταξης. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να επιβιώσουν κιόλα μετά την ε, αποχώρηση τους από την υπηρεσία. Εκεί όπου μπορούμε να έχουμε ένα περιθώριο για οικονομία, γιατί όχι. Μπορούμε να κάνουμε οικονομία παραδείγματι από τη Δερμηνία. Γιατί δεν χρειάζεται κάθε ομάδα εργασίας να έχει ε, μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Ε, κάθε χώρα και να βρούμε και κανένα δυο κάτω χώρες και δεν ξέρω τι που δεν έχουν και τόσο μεγάλο πληθυσμό ε, στη γλώσσα τους ε, Ολλανδοί, Δανείοι και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να μεταφράζονται τα έγγραφα σε κάθε γλώσσα. Γιατί να μεταφράζονται. Από εκεί μπορούμε να κάνουμε οικονομίες. Επίσης είμαι διατεθειμένη ε, τις οικονομίες αυτές να τις δεχθώ εφόσον όμως είναι λογικές, ορθολογικές. Σε κόστος από τα κτίρια ενδεχομένως, από το προσωπικό, ναι, αλλά σε ποιες θέσεις, σε ποιες βαθμίδες κτλ. Με τρόπο συνεπή και λογικό. Αυτό που δεν δέχομαι είναι εδώ να παίζει παιχνιδάκια το Συμβούλιο εις βάρος μας και μάλιστα να, να διώχνει και μάλιστα να, φέρνει εδώ πέρα υπαλλήλου, δημόσιου υπαλλήλου που καλά-καλά δεν ξέρουν μια ξένη γλώσσα να μιλήσουν, βρίσκονται σε κάποιο Βερολίνο ή σε κάποια Βόνη ή σε κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία και έρχονται εδώ να ενημερώσουν και να ε, λάβουν αποφάσει ενώ καλά-καλά δεν ξέρουν τι του συμβαίνει. Και με, με μέσο επίπεδο γνώσεων και κατάρτισης πολύ χαμηλό, αλλά πολύ υψηλό επίπεδο φθόνου εις βάρους των ευρωϊπαλλήλων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν σωστά, πρέπει να συζητήσουμε που μπορούμε να βρούμε περιθώριο για εξοικονόμηση πόρων, διοικητικό, διοικητική εξοικονόμηση κτλ. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω, ιδιαίτερω για κάποια κράτη όπω η Βρετανία που προσπαθούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι τη αμάυρωση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην ε, εγκρίνω το, ε, τα, κονδύλια για τα διεθνωτικά ταμεία μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Δεν με νοιάζει και εδώ σε 12 μήνε δεν εγκρίνουμε. Α μην έχει η Γαλλία την, ε, τα, τα, τα κονδύλια για τη γεωργία. Α μην πληρώσει. Α μην πληρωθούν οι επιδοτήσει και ό,τι χρειάζεται. Α ορίσουμε λοιπόν εμεί ποιοι είναι οι όροι του παιχνιδιού. Και ξέρω πολύ καλά ότι η Επιτροπή και ο κύριο Μπαρόσο και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερω. Ε, είναι στο πλευρό μας, αλλά εν πάση περιπτώσει ας συζητήσουμε και ας προαγάγουμε λίγο περισσότερο το ζήτημα της αιτιακής σχέσης δεν μπορούμε να λέμε ότι πάλι υπάλληλοι είναι όλοι ε, άχρηστοι, όλοι χαραμοφάιδες και ούτε καθεξής. Εάν θέλετε να δουλεύει το σύστημα, εάν θέλετε να έχουμε αποτελέσματα, τότε θα συστήσουμε όλοι λογικά. Διαφορετικά, εάν θέλει το καθένα να προβάλλει το δικό του θεματάκι και να το παίζει όπως το θέλει για, για την ε, προβολή του, τότε δεν θα είμαστε εμείς μέρος αυτού του παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή θέλει να λάβει τον λόγο, παρακαλώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω σε αυτό το στάδιο ότι η Επιτροπή ανησυχεί με τη μεγάλη καθυστέρηση αυτής της διαδικασίας. Αυτό οδηγεί μεγάλη ανησυχία και αστάθεια στο προσωπικό και στα θεσμικά όργανα. Η πρότασή μας για την τροποποίηση υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού βρίσκεται επιτάπητος εδώ και ένα χρόνο. Και η έκθεση Ροντ Μπέρεντ έχει εγκριθεί από εσάς οκτώ μήνες πριν. Γι' αυτό ας αρχίσουν οι τριμερείς διάλογοι και θα πρέπει αυτό να γίνει εντάχει και με σπουδή. Γιατί ε, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων από αυτή την καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ. Δύο από τους τρεις είναι στο, σε stand-by λοιπόν. Να δούμε ο τρίτος θα κάνει. Καλώς. Αφήνουμε το σημείο αυτό προς το παρόν για να περάσουμε στην παρουσίαση του Κέντρου Πολιτικής για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Κυρία Κράμερ, κύριε Ντερόι, ποιος θα ξεκινήσει. Ποιος θα κάνει την παρουσίαση.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 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω αυτή την παρουσίαση της μελέτης μας. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να το κάνω. Η αναθέσατε, μας αναθέσατε την εργασία αυτή. Είμαστε εμπειρογνώμονες από την Ολλανδία και ε, συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες από άλλα κράτη-μέλη. Οι κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου είναι σημαντικοί. Οποτεδήποτε υπάρχουν συμβατικές διεθνείς ρυθμίσεις, όπου υπάρχουν διασυνοριακές ε, συμβάσεις. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ρυθμίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους και γενικότερα σε, στα πλαίσια διεθνών συμβάσεων όπως τη Σύμβαση της Χάγης για το Διεθνές ε, Ιδιωτικό Δίκαιο. Ε, μετά τη συνθήκη του Άμστερνταμ το 1999 και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ουσιαστικές εξουσίες στον τομέα του διεθνου, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο νομοθεσίας έκτοτε και προφανές δεν λαμβάνεται υπόψη ε, ο κάθε περίπτωση υπάρχουν κενά. Δουλειά μας λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι να διαπιστώσουμε πού υπάρχουν αυτά τα κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία και ποιες είναι οι προσθήκες που απαιτούνται. Επιπλέον ασχοληθήκαμε με το θέμα εάν πέρα από τα μέσα που υπάρχουν τώρα θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο διαρθρωμένη και συνεκτική νομοθεσία. Σκοπός, το πεδίο εφαρμογή της μελέτης αφορά την διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και τους κανόνες αναγνώρισης και εφαρμογής και ε, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία αφήσαμε εκτός του πεδίου της μελέτης μας. Στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, και αυτό είναι σημαντικό και αξίζει να σημειωθεί, ε, παρότι ο τομέας είναι πολύ τεχνικός και παρόλο που η νομοθεσία είναι τεχνικής φύσεως, είναι πολύ σημαντικό σημαντικός ο τομέας αυτός για τους πολίτες και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο είναι σημαντικό για την λειτουργία της, της αγοράς ας πούμε στο εμπόριο. Επίσης υποστηρίζει την ελεύθερη διακίνηση ατόμων και επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί είναι και αυτοί ε, σημαντικοί για την ε, ενίσχυση του ε, ευρωπαϊκού ε, ε, χώρου οι κανόνε για το εφαρμοστέο δίκαιο είναι και αυτοί σημαντικοί γιατί θα πρέπει κάθε ευρωπαϊκό δικαστήριο να εφαρμόζει το ίδιο δίκαιο. Η ουσία του νόμου μπορεί να διαφέρει αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα προσφέρουν την ίδια ουσία, το ίδιο ουσιαστικό δίκαιο. Οι κανόνε επίση είναι σημαντικοί για τον ευρωπαϊκό νομικό χώρο. Δηλαδή να υπάρχει εγγύηση ότι ένα νομικό έγγραφο που συντάσσεται σε ένα κράτος μέλος θα αναγνωρίζεται σε άλλο κράτος μέλος και ότι μια δικαστική απόφαση που... Ε, λαμβάνεται σε, μια, σε ένα κράτος μέλος θα μπορεί να ε, εφαρμοστεί σε άλλο κράτος μέλος και αυτό ε, διευκολύνει τους πολίτες, τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Έτσι λοιπόν οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ε, αν εναρμονιστούν θα μπορούν να βοηθήσουν στην ευρωπαϊκή υπηκότητα. Τώρα όσον αφορά το πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς είναι σημαντική για τα δικαστήρια που πρέπει να εφαρμοστούν. Είναι επίσης σημαντική για άλλους χώρους, ας πούμε για τους συμβολιογράφους και τους δικηγόρους. Να σας δώσω ας πούμε κάποιες, ε, κάποια παραδείγματα. Ας πούμε δύο συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων σε διάφορα, διαφορετικά κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό αυτά, αυτοί να γνωρίζουν ποιο, που, ε, σε ποια δικαστήρια θα προσφύγουν και ποια ε, νομοθεσία ισχύει κάποιος που προσπαθεί να αποκτήσει αγαθά σε, κάποια, σε άλλο κράτος μέλος είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ας πάρουμε κάτι άλλο, μια παράνομη πράξη, ας πούμε, μια παραβίαση των ιδιωτικών δικαιωμάτων, παραβίαση των δικαιωμάτων προσωπικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια πρέπει να αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό με ομοιόμορφο τρόπο και να εφαρμόζουν το ίδιο δίκαιο. και επίσης πρέπει ε, να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όσον αφορά τις, ε, την αποκατάσταση. Στα περισσότερα κράτη-μέλη ε, η ονοματοδοσία γίνεται από το όνομα του πατέρα αλλά σε κάποια άλλα μπορεί να πάρει του πατέρα ή της μητέρας ενώ σε άλλα κράτη-μέλη η παράδοση λέει ότι παίρνουν το συνδυασμό πατρός και μητρός. Είναι λοιπόν σημαντικό αν θέλεις να έχεις ευρωπαϊκή υπηκότητα, οι διάφοροι κανόνες να γνωρίζονται αμοιβαία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καθώς συνεχίζεται η ζωή και καθώς παντρευόμαστε, χωρίζουμε, χρειαζόμαστε διατροφή για τα παιδιά, πρέπει να ισχύουν ομοιόμορφοι κανόνες, κυρίως λόγω της αυξημένη κινητικότητας. Οι άνθρωποι μετακινούνται από χώρα σε χώρα, πρέπει να γνωρίζουν, να είναι, εξασφαλισμένο, θα είναι αναγνωρισμένα τα δικαιώματά του. Να προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το εφιστάμενο πλαίσιο ε, τι κανόνες υπάρχουν. Είναι 13 διαφορετικοί κανονισμοί και δύο οδηγίε, και υπάρχουν και ε, ε, η εναρμόνιση πολλών από αυτών που εξακολουθούν να εκκρεμούν. Και ε, υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες για τους οργανισμούς και τους καταναλωτές, ας πούμε. Έχουμε καταλήξει ότι όλοι αυτοί οι κανόνες και η δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό είναι σημαντική. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην νομοθεσία και μάλιστα σημαντικά κενά. Και επειδή υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για τομείς όπως ε, το, το διαζύγιο και η διατροφή κλπ. Κάποιοι κανόνες ε, επαναλαμβάνονται. Υπάρχουν δηλαδή κανόνες που καθορίζονται από διαφορετικά μέσα και αυτό συνεπάγεται επιπλέον νομοθετική προσπάθεια. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ότι στο οικογενειακό δίκαιο υπάρχουν περιορισμοί. Ας πούμε η, η ομοφωνία που απαιτείται. Και στο παρελθόν, όσον αφορά το αφορμαστέο δίκαιο στην περίπτωση του διαδιζυγίου, αυτό δεν μπορούσε να συμβεί πάντοτε, δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό όσον αφορά τον εντοπισμό των ε, κενών που υπάρχουν στην νομοθεσία κοιτάξαμε το πεδίο εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων και τα αναλύσαμε. Επίσης κάναμε μια συστηματική ανάλυση δυνάμει των βασικών αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε σχέση με την εθνική νομοθεσία και με την ε, διεθνή κωδικοποίηση του ιδιωτικού διεθνούς όπως επίση και το υφιστάμενο συμβατικό δίκαιο και εντοπίσαμε τριών ειδών κενά. Πρώτον, το είδος που προκύπτει από τις Βρυξέλλες ας πούμε, όπου η νομοθεσία περιορίζεται Ε, ε, διέπεται από γενικές αρχές και μετά υπάρχουν σημαντικές ε, εξαιρέσεις, υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους ισχύουν οι διεθνείς συμβάσεις και μετά μπορεί να υπάρχει και συμβιβασμός. Και το πιο σημαντικό, μελετήσαμε τη συστηματική ανάλυση για τον εντοπισμό των κενών του συστήματος και διαπιστώθηκε ότι κάποιοι τομείς δεν ρυθμίζονται καθόλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι σήμερα. Και τα σημαντικά αυτά κενά αφορούν το δίκαιο των ακινήτων, των περιουσιακών στοιχείων τα καταπιστεύματα τους, ε, της και τα νομικά πρόσωπα και τα πρακτορία. Επίσης οι κανόνες ε, ε, διατησίας ας πούμε και αποκατάστασης. Ξέρω ότι από αυτού ισχύουν διεθνείς κανόνες, αλλά θα μπορούσαμε ίσως να προχωρήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτό το πεδίο. Έχει συζητηθεί εκτεταμένα διεθνώς η συλλογική αποκατάσταση. Είναι ένα σημαντικό ε, διαδικαστικό μέσο. Στον τομέα του οικογενειακού δικαίου έχουμε εντοπίσει τα εξή κενά. Στον τομέα του γάμου. Το εφαρμοστέο δίκαιο και η αναγνώριση των, για την αναγνώριση των γάμων ας πούμε. Υπάρχουν ε, ε εδώ κενά και όσον αφορά τις καταχωρημένες ε, σχέσεις. Έχουμε εντοπίσει κενό όσον αφορά τα ονόματα, κυρίως τα ονόματα των νομικών προσώπων. Ούτε η οθεσία έχει καλυφθεί, ούτε η γονική σχέση ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προστασία των πιο αδύναμων ενηλίκων είναι άλλος τομέας Όλα αυτά τα κενά έχουν σημαντικέ συνέπειε στην ελεύθερη διακίνηση ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θεωρούμε σημαντικό είναι ότι σε κάποιου από αυτού του τομεί υπάρχουν ε, ε, αποτελέσματα ε, που προέρχονται από τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές. Σε κάποιους από αυτούς τους τομείς, όπως ας πούμε στα ονόματα και στο δίκαιο των νομικών προσώπων υπάρχουν ε, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ευρωπαϊκή υπηκότητα και την ελεύθερη διακίνηση των ε, ατόμων, αλλά δεν έχει δοθεί επαρκής προσοχή στα, ε, στις πτυχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και πολλά πράγματα δεν έχουν κωδικοποιηθεί ακόμα. Σημαντικά θέματα για προσμελέτη, αν θέλουμε να καλύψουμε τα υφιστάμενα κενά ή να υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο ή το ιδιωτικό διεθνές να δούμε ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι. Οι εμπλεκόμενοι είναι αυτοί στους οποίους αναφερθήκαμε προηγουμένως. Οι Ευρωπαίοι ε, πολίτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και οι δικηγόροι και άλλα νομικά επαγγέλματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί ε, έχουν συμφέρον ε, να υπάρχει ένα διαρθρωμένο και συνεκτικό ε, σύστημα τέτοιου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορεί να πέσει, παίξει σημαντικό ρόλο και να επιφέρει μεγαλύτερη πρόοδο από ότι η διεθνή νομοθεσία, ας πούμε, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάρης κτλ. Αυτό που μπορεί να γίνει εδώ είναι δύο πράγματα. Είτε να υπάρξει σταδιακή εναρμόνιση για να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά ή να προσπαθούμε να κάνουμε μια πιο ε, διαδομημένη κωδικοποίηση ε, στην νομοθετική τεχνική. Ε, όμως πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στο οικογενειακό δίκαιο. Εκεί υπάρχουν τα περισσότερα κενά. Αλλά βεβαίως υπάρχει κυρίως η αρχή της ομοφωνίας. Εδώ μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί τεχνική της ενισχυμένης συνεργασίας. Και στο εφαρμοστό δίκαιο στην περίπτωση των διαζυγίων αυτό είναι σημαντικό. Ξέρω ότι έχει γίνει κάτι σε σχέση με τον βάση του κανόνα 3, αλλά ε, τίνει να χαθεί αυτή η τεχνική και δημιουργείται μάλλον περισσότερος κατακαιρματισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως και μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Έτσι λοιπόν το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί, να δούμε αν είναι επιθυμητό, τι έχουμε επιτύχει, τι θέλουμε να επιτύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν αυτό να είναι ένας τρόπος αποκατάστασης, η τελευταία δυνατότητα. Ένα άλλο θέμα είναι αν θα ήταν δυνατό σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα να υπάρξει ευρωπαϊκή κωδικοποίηση του ιδιωτικού διεθνές, έναν ευρωπαϊ... ευρωπαϊκός κώδικας αυτό που κάναμε με τους εμπειρογνώμονες των άλλων χωρών είναι ότι είπαμε ότι ίσως ένα ενιαίο ε, μέσο θα ήταν ίσως καλύτερο γιατί θα υπήρχε λιγότερος κατακαιρματισμός και αυτό σημαίνει ότι η καδικοποίηση ε, υπό την έννοια του ε, αστικού δικαίου θα ήταν πιο συστηματική θα, έκανε, θα αύξανε τη διαφάνεια του νόμου και θα βοηθούσε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για αυτούς που την χρειάζονται. Όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα που προέκυψε στη συζήτησή μας με τους ξένους εμπειρογνώμονες ότι αν εντός Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε όλη την ίδια αντίληψη του TST κωδικοποίηση. Ας πούμε οι χώρες του ε, κοινοδικαίου, του common law, δεν έχουν την ίδια ε, έννοια της κωδικοποίησης όπως οι χώρες του αστικού δικαίου και στις ευρωπαϊκές νομοθετικές τεχνικές ο όρος κωδικοποίηση έχει δική του έννοια και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τώρα, πρέπει να ε, συμφωνήσουμε ότι όλοι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Επίση, στα κράτη-μέλη, ακόμα και στις, στους ακαδημαϊκούς κύκλους, υπάρχει πολύ θετική ε, υποδοχή στην άποψη να υπάρχουν ε, ευρωπαϊκοί κώδικες. Ας πούμε, η, μια τέτοια συζήτηση γίνεται στη Γερμανία και τη Γαλλία. Αλλά δεν ισχύει αυτό σε άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο στους ακαδημαϊκούς κύκλους, αλλά και στις κυβερνήσεις. Δεν αισθάνονται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Οι του ιδιωτικού διεθνούς ας πούμε, όπως ε, η εφαρμογή του ξένου δικαίου ή των θεμάτων δημόσιας τάξης δεν έχουν αποκρισταλωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο και υπάρχουν τα κενά που ανέφερα προηγουμένως και τα οποία υπάρχουν οι χώροι που δεν, που δεν ρυθμίζονται καθόλου. Ίσως όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πριν ε, σκεφτούμε για έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε διαφορετικό ουσιαστικό δίκαιο στο θέμα ας πούμε των σχέσεων μεταξύ συντρόφων. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές και αυτό πρέπει να το λύσουμε πριν αρχίσουμε καν να διανοούμε στην κωδικοποίηση. Ε, κλείδι καταλήξαμε ότι μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει έμφαση στο να καλύψει τα υφιστάμενα κενά επί στον τομέα που ανέφερα. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε μια βαθμιαία εναρμόνιση των διαφόρων μέσων όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Μακροπρόθεσμα όμως, δηλαδή σε διάστημα 15 ετών θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την εδραίωση της ε, ε, ισχύουσας νομοθεσίας αφού θα έχει γίνει κάποια πρόοδος σε όλους τους τομείς και θα μπορέσει να συνταχθεί ένας ευρωπαϊκός κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, θέλετε να προσθέσετε κάτι κι εσείς. Όχι θα αρκεστώ σε αυτά που είπε η συνάδελφος. Καλώ, τότε υπάρχουν ερωτήσει, Κυρία Λίχτινμπέργκερ. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με την ανάλυση σας. Το μόνο μου ερώτημα είναι το εξής. Εάν έχουμε εδώ ενισχυμένη συνεργασία εν γέννη, Τότε μήπω επιδεινώνεται η κατάσταση, μήπω ε, την καθιστούμε πιο δύσκολη. Διότι εν τέλει, ανάλογα με το κράτος προελεύσεως, πάλι έχουμε διαφορετικές ρυθμίσεις μέσα στον ευρωπαϊκό, χώρο. Και άρα για λόγους ασφάλειας και σαφήνειας του δικαίου, θα έπρεπε ίσως να δοθεί μια διαφορετική λύση. Έχω κάποιες επιφυλάξεις λοιπόν. Αντιλαμβάνομαι γιατί κανείς καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα, γιατί όλα τα θέματα αυτά κρίνονται με τρόπο αρκετά, αντιμετωπίζονται με τρόπο αρκετά συγκινησιακό στα κράτη-μέλη και για ορισμένα. Για ορισμένα ζητήματα δεν μπορούμε να προσμένουμε ξαφνικά να ξυπνήσουν μια μέρα και να αντιμετωπίσουν με απλή λογική να έμπλεει ε, ορθολογικού πνεύματος να ε, δώσουν διαφορετικές λύσεις. Εδώ μιλούμε για συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένα μειονεκτήματα στα οποία ε, τα οποία αντιμετωπίζουν, ε, τα, ε, από, τα οποία πλήττονται σε περίπτωση που βρίσκονται σε υπερσυνοριακές σχέσεις. Αλλά επισημαίνω η ενισχυμένη συνεργασία είναι πάνω από το, το πρόβλημα εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ας ακούσουμε λοιπόν και άλλους. Η κυρία Τάιν. Έχω μια ερώτηση. Εάν αυτό το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο του Δυτικού Διεθνούς Δικαίου ε, έχει κάποια νομική βάση συγκεκριμένη ή μήπως είναι και αυτή αμφιλεγόμενη όπως με το Γενικό Εμπορικό Δίκαιο. Δεν έχω πρόχειρη απάντηση. Δεύτερη ερώτηση μας. Ε, μιλήσατε για πολλά, πολλά κενά. Ποια θα ήταν ίσως τα πιο κατεπήγοντα. Δεν ξέρω αν το ζήτημα της ονοματοδοσίας είναι το πιο επίγον, αλλά ή το, το ε, δίκαιο της υιοθεσίας, ίσως κάποια άλλα θέματα τα οποία όμως έχετε το ως πιο επίγοντα, να μπορούσαν να πάρουν προτεραιότητα. Επίσης το θέμα της ενισχυμένης συνεργασίας. Όσον αφορά την αναρμόνιση έχουμε δει πολλές δυσκολίες και ιδιαίτερα στο οικογενειακό δίκαιο βλέπουμε ότι έχουμε σημαντικές αποκλήσεις μεταξύ μας και στο διεθνές, ε, στο δυτικό διεθνέ δίκαιο ιδιαίτερα εντοπίζεται η διαφορά σε σχέση με το common law, με το δίκαιο το αγγλοσαξονικό. Επομένω, πρέπει να κοιτάμε κάθε φορά ποιο έχει προχωρήσει μέχρι ποιου σημείου, ποια κράτη έχουν δώσει κοινέ λύσει σε ποια θέματα και να κάνουμε έτσι ένα μακροσκελή κατάλογο στον οποίο θα μπορούμε να παραπέμπουμε κατά περίπτωση. Είναι μια Ευρώπη αλακάρτου ουσιαστικά που δεν την προτιμώ αλλά αν δούμε ο κανονισμός περί διαζυγίου περί πόσο δυσκολίες γέννησε, πόσο πολύ καθυστέρησε και τελικά τι αποτελέσματα έδωσε. Ε, είναι νομίζω δύσκολο και με δεδομένες ενδεχόμενες ε, ε, διευρύνσεις στο μέλλον με πάνω από 25 μέλη, εν πάση περιπτώσει, θα είναι δύσκολο να βρούμε λύσει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σιμάνσκι. Ένα σχόλιο έχω ε, αποκλειστικά να υποβάλω. Στο εγγύς μέλλον δεν μπορώ να φανταστώ να έχουμε έναν ε, Ευρωπαϊκό Κώδικα για το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο. Αυτός είναι βεβαίως ο απότερος στόχος, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε βήμα προς βήμα με όλα τα στοιχεία του διεθνούς δικαίου που προπετούνται. Γιατί, εάν λάβουμε υπόψη το μέλημα των πολιτών, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. να προβούμε σε μία ιεράρχηση. Βεβαίως το πλαίσιο Βρυξέλλες 1 δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό, αλλά πρόσφατα κάναμε ένα σημαντικό βήμα που δείχνει ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατόν. Όταν φτάσουμε σε, ένα, σε μια καθαρά ε, ομοσπονδιακή δομή, κάτι το οποίο προσωπικά θα μου ήταν ιδιαίτερα αρεστό, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την εναρμόνιση του νόμου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονές μας, δεν πιστεύετε ότι τα σημεία του νόμου που ενέχουν αυτό το χάσμα όπως το έχετε ορίσει σκοπίμως ε, μένουν εκτός εμβέλειας ε, όλων των διευθετήσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμφιλιώσουμε τις εθνικές ένομες τάξεις. Δηλαδή στη δική μου χώρα τα καταπιστεύματα δεν υπάρχουν με αυτή τη μορφή που τα εννοείτε εσείς. Και αυτά τα λεπτά ζητήματα που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκαιο και με το δίκαιο της διαδοχής καθιστούν πολύ δύσκολη τη σύγκληση μεταξύ εσωτερικών ένωμων τάξεων. Επίσης, ο εθνικός νομοθέτης είχε λόγο συμμετοχής ή opt-out. Και ό,τι προέρχεται από τις Βρυξέλλες ίσως φαίνεται ότι είναι κάποιο δόγμα. Σε σχέση τώρα με το δίκαιο της ιδιοκτησίας και με το ενοχικό δίκαιο, νομίζω ότι τα συστοιχίσατε και δεν νομίζω ότι συνυπάρχουν υπό την ίδια κεφαλίδα. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεφτενμπέργκερ. Μια παρατήρηση Δικτάτα από τις Βρυξέλλες, εντολές από τις Βρυξέλλες λέτε, αλλά που φαίνεται παράξενη αυτή η λέξη, γιατί όταν αποφασίζετε κάτι αποφασίζετε από κυβερνήσεις. Επομένως τι είναι αυτό, διαταγές, εντολές από τις Βρυξέλλες. Καλώς κυρία Κράμερ, για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και συμφωνώ απολύτως κυρία Λιχνιμπέργκερ στα όσα είπατε για την ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει όσο δυνατόν να την αποφεύγουμε. Θα μπορούσαμε βεβαίω να πούμε όπως έγινε με τη Ρώμη 3. 15 κρατη έχουν προχωρήσει και μπορούν να, να πάνε μαζί. Και έτσι διευκολύνεται η κατάσταση για ορισμένους. Ή αλλιώς κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε περισσότερο κατακαιρματισμό στην νομοθεσία. Ε, έτσι λοιπόν το θέμα δεν είναι τόσο τα 5, τα 10, τα 20 κράτη-μέλη που θέλουν να κάνουν κάτι. Είναι, το θέμα είναι να πιστούν όλοι να προχωρήσουν μαζί. Αυτή θα είναι η πραγματική πρόοδος. Για τη νομική βάση. Προσπάθησα να το υπογραμμίσω. Πρόκειται για το άρθρο 81 της συνθήκης, το οποίο αναφέρεται σε ειδική, ειδική ενσημένη συνεργασία για την εναρμόνιση. Δεν έχει σημασία λοιπόν εκεί πέρα το θέμα, όσο η αρμοδιότητα, περιορισμένη αρμοδιότητα για όλα αυτά τα θέματα, για την αναγνώριση, την εκτελεστότητα, όλα αυτά τα θέματα που έχουν διασυνοριακές συνέπειες. Η νομική βάση μπορεί να μην επιβάλλει απαραίτητα σε περίπτωση θεμάτων που αφορούν τα παιδιά στο οικογενειακό δίκαιο την ομοφωνία αλλά μπορεί να ε, περάσει, από κάποιο κράτος, ε, μπορεί να περάσει κάποιο κράτος μέλος τη δυνατότητα του αυτοαποκλεισμού, της αυτοεξαίρεσης, του opt-out, παραδείγματι, ή αντίστροφα του opt-in. Ε, αυτά όλα είναι δυσκολίες. Μετά υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το οικογενειακό δίκαιο λόγω των πολύ διαφορετικών διατάξεων ουσιαστικού δικαίου αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω θα ξεκινούσα καλύτερα από το περιουσιακό ή από τα θέματα της ε, κυριότητας και τα λοιπά, τα θέματα τα ιδιοκτησιακά, τα οποία και λόγω της οικονομικής κρίσης θα έχουν και περισσότερη απήχηση. Η δε νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, την ελευθερία εγκατάστασης κτλ ήδη έχει δώσει τόσες πολλές ρυθμίσεις, αν όχι ρητές με μέσω του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου πάντως μπορεί να δοθούν ε, απαντήσεις και έτσι δεν νομίζω ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα ιδιαίτερο. Στο οικογενειακό δίκαιο, όπως είπα, είναι πολύ διαφορετικοί οι ισχύοντες κανόνες. για την σύναψη είτε ελεύθερη σχέση, είτε καταχωρημένη σχέση, είτε ε, γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου, ε, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συζύγων, ως προς τις συνέπειες από την αποκτήση τέκνων, όλα αυτά τα θέματα, τα οποία με την μέθοδο της αμοιβαίας αναγνώριση, όταν δηλαδή κάποιος ε, που έχει το καθεστώς αυτό πηγαίνει σε ένα άλλο κράτος μέλος πρέπει να είναι ή μη τι άλλο ανεγνωρισμένη έστω και αν δεν μπορεί το κράτος υποδοχής να δημιουργήσει το θεσμό αυτόν τουλάχιστον πρέπει να τον αναγνωρίζει, να αναγνωρίζει την ε, ένομη σχέση όπως προέρχεται από το κράτος, ε, το προηγούμενο κράτος εγκατάστασης. Εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο εγχείρημα, ένα μεγάλο εγχειρίδιο ή ένα κώδικα του Δυτικού διεθνούς δικαίου δεν μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα έχουμε σύντομα. Αλλά για τα θέματα αυτά τα οποία βεβαίως σε ένα βαθμό ε, ξεπερνούν τα όρια τις αρμοδιότητες, αλλά πρέπει να πω ότι και πριν από 10 χρόνια ήταν άλλες αρμοδιότητες και σε 10 χρόνια πάλι διαφορετικές θα είναι οι αρμοδιότητες. Άρα καλό θα είναι να επιδιώκουμε πάντοτε την ε, προσέγγιση, έστω και αν δεν έχουμε πάντα σαφή εικόνα. Νομίζω ότι για θέματα νομικών προσώπων λοιπά μπορούμε να βρούμε λύσεις χωρίς να αγγίξουμε το εσωτερικό δίκαιο στην περίπτωση των υπερσυναριακών ε, ένομων σχέσεων, εκεί που υπησέρχονται διαφορετικά ε, διαφορετικές έρωμες τάξεις, να βρούμε μια λύση που θα, αποτελεί, θα δίνει γέφυρα σε βάση περιπτώσει για τον πολίτη. Ο πρόεδρος ευχαριστώ πολύ. Ήταν ε, πολύ σημαντική αυτή η έκθεση που μας παρουσιάσατε και που βεβαίως δίνει νέα πνοή στις συζητήσεις μας. Ας δούμε τώρα το σημείο 23 και μετά θα πάμε στην ε, συνεδρίαση και των θυρών. Η κυρία Λιχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε το θέμα λοιπόν των προσωπικών δεδομένων και τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε είναι ζητήματα εξωτερικ... όχι εξωτερικών ε, αρμοδιοτήτων, αλλά πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα ως προς την διάρκεια που ε, ως προς τη διάρκεια των διαδικασιών εδώ υπάρχει μια αύξηση της διάρκειας στις ε, προδικαστικές αποφάσεις και σε ορισμένα ένδικα μέσα ή βοηθήματα σχετικά μεγάλη δυστυχώς, άρα υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο βελτίωσης. Κοίταξα εδώ ότι είδου ε, αποφάσεις ε, έχουν εκδοθεί. Και επίσης δεν θέλω να πω ότι εάν λειτουργήσει, ε, εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία μπορούμε να περιμένουμε καλά αποτελέσματα χωρίς πολλές καθυστερήσεις. Μπορούμε να μειώσουμε αυτό που ονομάζεται χειρόγραφη διαδικασία και να περάσουμε στις νέες τεχνολογίες, σε παραδείγματι, που θα επιταχύνουν πολύ την παραγωγή αποτελέσματος. Η διοικητική τάξη βεβαίως μας βρίσκει σύμφωνο, την υποστηρίζει και το δικαστήριο το 2013 και όχι το 1913 όπως πήγαν από αρχικά χρειάζονται κάποιοι, χρειάζεται να εξεταστούν και κάποια διαρθωτικά μέτρα πάντως ιδιαίτερα υπογραμμίζουμε ότι χρειάζεται να διοριστούν και επιπρόσθετοι δικαστές. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει από καιρό. Όχι μόνο οι διατυπώσεις αλλά και η κατανομή ανακράτος μέλος ή κάποια κρατημέλη. Πάντως ελπίζω να βρεθεί σύντομα η λύση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λιχτινμπέρκερ. Υπάρχουν ε, παρατηρήσεις. Όχι, ο Ταντέους, έλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάχει, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όσα προείπε η Εύα. Αυτή η μεταρρύθμιση λειτουργίας του δικαστηρίου είναι ύψης της σημασίας. Βέβαια σήμερα η οικονομική κατάσταση δυσχεραίνει αυτό το έργο, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει το δικαστήριο να προβεί σε αυτή τη μεταρρύθμιση και σας υποστηρίζουμε πλήρως. Ευχαριστώ προθεσμία. Τίποτα άλλο κύριε όχι προθεσμία. 20 Τώρα προχωρούμε σε συνεδρία κυκλισμένων των θυρών. Όποιος δεν έχει εδώ εργασία, παρακαλώ να αποχωρήσει. Διακόπτω για δύο λεπτά τη συνεδρίαση για να γίνει και η σχετική προσαρμογή, να σταματήσει το web streaming κτλ.